almost the, academic we call passed already. So... Σχεδόν πέρασε το ακαδημαϊκό τέταρτο, γι' αυτό θα αρχίσουμε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας μας, καθώς και τα μέλη της αντιπροσωπείας με τις χώρες μας ΡΕΚ, που είναι παρόντα στην συνεδρίαση, στη συζήτηση. Την κυρία Ρόιγ Γκρονζόν από την ύπατη αρμοστία των προστίγων και τον κύριο Πακέ, ο οποίος είναι ε, υπεύθυνο για θέματα τουρκικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε βεβαίως ε, τον κύριο Καμακτσί, ο οποίος είναι ο πρέσβης της Τουρκίας. Θα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μαρίζα Ματέη, που είναι πρόεδρος αντιπροσωπείας της χώρας Μασρέκ. Έχουμε δύο ερμηνεία σε επτά γλώσσες. Γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ελληνικά, ισπανικά και πορτογαλικά. Δεν υπάρχουν αλλαγέ στην ημερήσια διάταξη. Θεωρώ ότι εγκρίνεται. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω, να ενημερώσω τα μέλη των δύο για τις πρόσφατες εξελίξεις της αντιπροσωπείας μας, μας με την Τουρκία συζητούμε όλα τα θέματα που αφορούν τις ε, διακοινοβουλευτικές σχέσεις με την Τουρκία. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Μαρίζα Ματίας. Από την ε, συνάντηση που είχε γίνει στην Άγκυρα πριν από δύο χρόνια μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει άλλη συνεδρίαση. Θα γίνει μία τον Ιανουάριο του 2018 έγινε μια γενική συζήτηση επί αυτών των θεμάτων και ενημερωθήκαμε ότι ο κύριος Ισμαέλ Καραγγέλ είναι συνεισηγητής για τα θέματα που με απασχολούν εκ μέρους της Τουρκής Πρόκειται κατά την άποψή μου για μία ευκαιρία να ξαναρχίσουμε τον διάλογο. Θα καλέσουμε τον κύριο Καραγγέλ. Τον έχουμε ήδη καλέσει στην συνεδρίαση που κάναμε στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο. Συμμετείχε σε εργασίες μας και ανταλλάξαμε απόψεις. Είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση του Προεδρείου, το συντομότερο δυνατό, μας είπε ο κύριος Κάλαγκελ, ότι μια ε, συνεδρίαση του Προεδρείου θα πρέπει να γίνει το, στην Άγκυρα το Μάρτιο, συμφωνήσαμε και είπαμε ότι θα συζητήσουμε τις ε, λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ματίας για να κάνει τις εισαγωγικές παρατηρήσεις και τα σχόλιά της. Έχει το λόγο κυρία ματίς. Thank you. I'm going to speak in Portuguese. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν θα ήθελα να καταναλώσω το χρόνο μας με εισαγωγικέ παρατηρήσεις. Πιο σημαντικό είναι να ακούσουμε τους προσκεκλημένους και να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Μετά από την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αποφασίσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μία συνεδρίαση από κοινού μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών μας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες Σύριοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Τουρκία. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε το όλο θέμα, διότι από τα στοιχεία που έχουμε, ξέρουμε το 94% των προσφύγων της Συρίας ζουν εκτός καταβλισμών προσφύγων. Σε συνθήκες πραγματικά προκλητικές, με ελάχιστους πόρους. Και η πλειοψηφία μεταξύ των προσφύγων αυτή τη στιγμή ζει κάτω από δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Βρίσκονται κάτω από το κατόφλι της φτώχειας και σε άκρα ένδια βρίσκεται το 1 τέταρτο αυτών. δεν θα κάνουμε μαθήματα ηθικής τώρα για το πώς χειριζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους πρόβλης, αλλά επειδή έχει υπογραφεί η σχετική συμφωνία ένθεν και ένθεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, τίθενται πολλά θέματα τα οποία πραγματικά είναι πρόκληση στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Το Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τη σημερινή συζήτηση, να δούμε από την οπτική γωνία του διεθνούς δικαίου ποιοι είναι οι κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται και πώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν λοιπόν στη σε αυτή που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και κυρίως τους προσκεκλημένους μας οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά μας. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε την κυρία Ματίας. Mrs. Ε, head Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς θα ήθελα να σας παρουσιάσω γενικώ την κατάσταση των σύρων προσφύγων στην Τουρκία και τις ανησυχίε για την προστασία τους που μπορεί να έχουμε. Έχω προετοιμάσει μια παρουσίαση, κάποια αριθμητικά στοιχεία θα τα βλέπετε και στην οθόνη. ελπίζω να έρθει και ο πρέσβης ώστε να μπορέσει να συμπληρώσει ε, ίσως κάποια πράγματα που, θα, δεν θα πω εγώ. Θα ξεκινήσω όμως με κάποιες γενικές έτσι πληροφορίες. Η Τουρκία όντως είναι η μεγαλύτερη χώρα που φιλοξενεί πρόσφυγες στον κόσμο έχει ξεπεράσει το Πακιστάν και το Αφγανιστάν που ήταν παλαιότερα οι μεγαλύτερες χώρες με τις μεγαλύτερες ε, ε, ομάδες προσφύγων. Στην Τουρκία βρίσκονται αυτή τη στιγμή 3,4 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες ε, εθνικότητες και άλλοι άνθρωποι δηλαδή άλλων εθνικότητων που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας στην Ευρώπη. Στην Τουρκία αυτή είναι περίπου 300.000 από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Ιράν, τη Σομαλία και άλλες εθνικότητες. Όλοι νομίζω ξέρουμε ή θυμόμαστε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να έχει μια γεωγραφική, ένα ε, γεωγραφικό περιορισμό για την συνθήκη της Γενέβης και το καθεστώς του πρόσφυγα, οπότε η Τουρκία είναι συνυπογράφων μέρος της Σύμβασης της Γενέβης αλλά όχι στο πρωτόκολλο 67 που έχει διευρύνει την ε, αρχική στόχευση του προς όλο τον κόσμο και την προστασία των ε, προσφύγων. Η Τουρκία λοιπόν συμφωνεί να φιλοξενεί Ευρωπαίους ε, πρόσφυγες ή ετούντες άσυλο, αλλά όχι άλλους. Αυτό σημαίνει η ετουντες ασυλο αλλα οχι αλλους αυτο σημαινει γεωγραφικη γεωγραφικός περιορισμός. Βεβαίως από τα νούμερα που βλέπετε ήδη, η Τουρκία ήδη έχει ε, πρόσφυγες Σύρους, αλλά όχι στα πλαίσια της ε, ε Σύμβασης της Γενέβης, αλλά μέσω διεθνούς νομοθεσίας. Μετά την πρώτη μαζική άφηξη Σύρων προσφύγων στην Τουρκία, η κυβέρνηση υιοθέτησε δύο νομοθετικά κείμενα που είναι πολύ σημαντικά. Ένα έχει να κάνει με την νομοθεσία για τη διεθνή προστασία που ρυθμίζει το καθεστώς του πρόσφυγα για τους Ευρωπαίους ετούντες άσυλο και για μη Ευρωπαίους. Και άλλο ένα νομοθετικό κείμενο που είναι η προσωρινή προστασία που αφορά στους σύρους πρόσφυγες και τους δίνει de facto καθεστώς προστασίας. Προσωρινό έστω. Από τα 3,4 εκατομμύρια σύρων προσφύγων, τα δύο τρίτα είναι γυναίκες και παιδιά, όπως βλέπετε. Η μεγάλη πλειοψηφία ζουν σε αστικές περιοχές, λιγότεροι στην Ήπεθρο και κάποιοι άλλοι ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων, τα οποία βεβαίως διαχειρίζεται η κυβέρνηση που βρίσκονται όλα στα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας. Βλέπετε πού βρίσκονται κυρίως στην Τουρκία οι Σύριοι πρόσφυγες, η πλειοψηφία σε μεγάλα αστικά κέντρα, 500.000 στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, Άγκυρα, Σμύρνη, και μεγάλη πλειοψηφία των 3,4 ε, εκατομμυρίων στα ανατολικά σύνορα της χώρας. Βεβαίως ε, δεν είναι λίγες οι προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει η Τουρκία για να καλύψει την κατάσταση αυτή. Συνεχίζει βεβαίως από την αρχή να δείχνει ότι έχει δυνατότητα να υποδέχεται ε, και να καλύπτει τις ανάγκες των προσφύγων σε μεγάλους αριθμούς. Η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει την ε, κατοχή, την διευθυνσία πούμε, του προγράμματο αυτού και την διαχείριση της περιοχή και βεβαίω υπάρχουν και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που συνδράμουν στο πλαίσιο που έχει ορίσει η κυβέρνηση. Το νομοθετικό πλαίσιο και το ε, επιχειρησιακό πλαίσιο. Ο κανονισμός τώρα για την προσωρινή προστασία προσφέρει πρόσβαση στους σύρου σε δημόσιε υπηρεσίε, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και σε κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό ήταν πραγματικά με αρκετά προοδευτική προσέγγιση και αυξάνεται κάθε χρόνο. Σε σχέση τώρα με την εκπαίδευση, από φέτος υπάρχουν πάνω από 600.000 παιδιά στην ε, πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 17.000 φοιτητές που έχουν ε, περάσει στο πανεπιστήμιο. Βεβαίως μετά από τόσα χρόνια υποδοχής και φιλοξενίας και ένταξης προσφύγων και πρόσβασής τους στις δημόσιες υπηρεσίες, οι προκλήσεις είναι πολλές και βεβαίως ε, υπάρχει μεγάλη πίεση στις δημόσιες αυτές υπηρεσίες ακριβώς επειδή αυξάνεται και η ζήτηση στατιστικά. Και υπάρχουν και πολύ περιορισμένες δυνατότητες παροχής τέτοιων υπηρεσιών σε κάποιες περιοχές. Και αυτό σημαίνει πίεση όχι μόνο για τους ε, πρόσφυγες, αλλά και για τον πληθυσμό των ε, ντόπιων που ζει στις πόλεις αυτές. Αυξανόμενη λοιπόν η ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις στις ε, τοπικές υποδομές και στις δυνατότητες που έχουν οι τοπικές αρχές να αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη ζήτηση. Μετά. Υπάρχει μια διευρυμένη κατάσταση εκτοπιστέντων. Δεν μιλούμε μόνο για τις ε, πόλεις που φιλοξενούν ή τις χώρες που φιλοξενούν, τους πρόσφυγες οι οποίοι, και οι οποίες πιέζονται, αλλά και ο ίδιος ο πληθυσμός πιέζεται. Διαπιστώθηκε από κάποιες αρχικές αξιολογήσεις, εκτιμήσεις, ότι λίγο περίπου πριν από ένα χρόνο πάνω από 18% των Σύρων ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τροφή και το τονίζω αυτό γιατί πριν από ένα χρόνο ε, το ποσοστό θα ήταν ε, ψηλότερο. Ε, ένα χρόνο μετά έχουν, έχει αυξηθεί η πρόσβασή τους στην, ε, στις διάφορες υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες. Υπάρχει και το δίκτυ ασφαλείας. Φαντάζομαι ότι η Κομισιόν θα το σχολιάσει. Και βεβαίως αυτό έχει αντίκτυπο και, στην, και στον πληθυσμό. Οι Σύριοι πρόσφυγες πρέπει να βρουν μηχανισμούς αντιμετώπισης για να επιβιώσουν. Και αυτό σε πολλές περιοχές είναι δύσκολο. Υπάρχουν πολλοί ε, τροτές ε, ευαίσθητες οικογένειες που έχουν να αντιμετωπίσουν διαφόρων ειδών προβλήματα. Τώρα, τι επέτρεψε τη βελτίωση της κατάστασης. Η δυνατότητα των σύρων προσφύγων να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση. Και αυτό είναι, έγινε χάρη σε μια νέα νομοθεσία που ε, έγινε, υπήρξε το 2016. Όλοι οι, οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας μπορούν να κάνουν αίτηση για άδεια εργασίας και έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της Τουρκίας. Μεγάλες οι προσδοκίες από αυτό το νομοσχέδιο με την έγκριση αυτή της ε, πρόσβασης στην ε, αγορά εργασίας και υπολογίζεται ότι περίπου 26.000 άδειε εργασίας έχουν ήδη δοθεί σε σύρους που βρίσκονται στο καθεστώς προσωρινής προστασίας. Παρόλα αυτά, για να έχει κανείς πρόσβαση στην απασχόληση, υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Ας πούμε, το γλωσσικό εμπόδιο, κοινωνικά, διοικητικά εμπόδια, το ποσοστό ανεργίας που επηρεάζει πολύ και τους, πολύ περισσότερο τους Τούρκους από τους Σύρους. Τα τέλη που πρέπει να πληρώσουν οι εργοδότες και επίσης κάποια, κάποιες ποσοστώσεις που πρέπει να τηρούν οι εργοδότες για την απασχόληση ξένων ή σύρων πολιτών. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη να συνεχίσει η διεθνής κοινότητα να υποστηρίζει την εφαρμογή αυτών των κανόνων για τις άδειε εργασίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουν περισσότερη, επιτρέψουμε την πρόσβαση σε περισσότερους Σύρου πρόσφυγες στην αγορά εργασίας. Τα παιδιά τώρα. Προστασία. Μεγάλο ποσοστό ακόμη των παιδιών δεν έχουν εγγραφεί σε σχολεία. Άρα ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και πρέπει και αυτά να εξεύρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Πολλές φορές υποχρεούνται να δουλέψουν και γενικώ υποχρεούνται να αντιμετωπίσουν πολύ δύσκολε καταστάσει. πρόσβαση λοιπόν στην εκπαίδευση έχει αυξηθεί μεν, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών εξακολουθούν να μην έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μια γενική εικόνα τώρα του πώς δουλεύει η διεθνής κοινότητα στην Τουρκία. ...270 εταίροι. Όλοι δουλεύουμε κάτω από ένα γενικό πλαίσιο το σχέδιο για την ανταπόκριση και την ε, αντίσταση για τους πρόσφυγες με αξιολογήσεις των αναγκών, με, θε... με κοινούς στόχους για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, σε στενή βεβαίως συνεργασία και με συντονισμό από την τουρκική κυβέρνηση. Η σύνδεση μεταξύ ανθρωπιστικών ε, οργανώσεων ε, βοηθά στην κάλυψη των αναγκών και βεβαίως υπάρχουν και τα εθνικά σχετικά σχέδια. Το σχέδιο λοιπόν αυτό καλύπτει τις ανάγκες των προσφύγων που ζουν στα διάφορα στρατόπεδα ή στις, ε, στους αστικούς κόμβους και θέτει και κάποιες προτεραιότητες για την περίοδο 2018-2019 για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, υγειονομικών υπηρεσιών μέσω του εθνικού συστήματος της χώρας που φιλοξενεί τους πρόσφυγες, άμεση βοήθεια στα ευαίσθητα κομμάτια της κοινωνίας και στους σύρους και βεβαίως ε, παροχή προς ε, ευκαιριών για την ε, καλύτερη ευημερία των σύρων προσφύγων. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες. Μπορώ να σας πω και ποιες είναι οι προτεραιότητες της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για την ε, ανταπόκριση στην κατάσταση στην Τουρκία. Συνεχίσουμε βεβαίως να συνεργαζόμαστε με την ε, τουρκική κυβέρνηση για να προωθήσουμε την πρόσβαση και την παροχή προστασίας. Προωθούμε και προετοιμαζόμαστε για βιώσιμες λύσεις για, τις, ε, για τους πρόσφυγες. Επιστροφές στην χώρα προέλευσης, ένταξη στην χώρα υποδοχής ή μετεγκατάσταση σε μια τρίτη χώρα. Αυτέ είναι οι τρει βασικέ προτεραιότητε προ αυτό. Μετά, ενίσχυση τη πρόσβαση σε ποιοτικέ υπηρεσίε για του πρόσφυγε μέσω ε, των δημοσίων υπηρεσιών. Και τέλος, προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες που υπάρχουν. Βεβαίως μπορώ, αν θέλετε, να μπω και σε περισσότερες λεπτομέρειες ως προς αυτό. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρέσβη, τον κύριο Καϊμακτσί και θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Πακέ από το τμήμα για την Τουρκία και κατόπιν κύριε πρέσβη θα ολοκληρώσετε εσείς τη συζήτηση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη. Ε, αγαπητοί συνάδελφε από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για τους πρόσφυγες. Θα ήθελα σύντομα να σας αναφέρω την προοπτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Φυσικά, συγκεκριμένο στοιχείο είναι η συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την Τουρκία ε, στο πλαίσιο της ε, δήλωσης του Μαρτίου του 2016 Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που πιστεύουμε ότι συνεχίζει να ε, επιφέρει καλά αποτελέσματα. Ήδη έχουμε πολύ λιγότερα μοιραία περιστατικά ανθρώπων που προσπαθούν να περάσουν τη Μεσόγειο. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εφαρμογή αυτής της δήλωσης και η επόμενη έκθεση θα αποτελέσει τμήμα της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για, την, για το θεματολόγιο της μετανάστευσης. Είναι σημαντικό πάντα να τονίσουμε, όπως ε, έκανε και η Άννα Μπελρόικ, είναι πάντα σημαντικό να αναφέρουμε τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει από πλευράς των τουρκικών αρχών, ε, που υποδέχονται 3,4 εκατομμύρια σύρων προσφύγων και 300.000 πρόσφυγες από άλλες χώρες. Παρακολουθούμε το σύστημα προστασίας που εφαρμόζει η Τουρκία και η αξιολόγησή μας θα συμπεριληφθεί στην ετήσια έκθεση για την Τουρκία που θα δημοσιευτεί μέσα Απριλίου. Θα ήθελα όμως να τονίσουμε τώρα τη δουλειά που κάνουμε από κοινού. Διότι προφανώς σημαντικό στοιχείο της δήλωσης είναι η διάθεση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίξει τις προσπάθειες της Τουρκίας όσον αφορά την υποδοχή αυτού του πολύ μεγάλου αριθμού προσφύγων. Σήμερα γενικά βρίσκομαι σε πολύ καλή θέση, διότι μπορώ να σας ανακοινώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει τους πόρους αυτούς εντός των προθεσμιών που ε, έληξαν στο τέλος ε, της περσινής χρονιάς ε, και σε περίπτωση που δεν γινόταν έγκαιρη απορρόφηση θα χάνονταν ε, αυτές οι δυνατότητες χρηματοδότησης. Τα καταφέραμε όμως και μάλλον είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε τόσο σύντομα στην ιστορία μας. 70 προγράμματα ήδη έχουν ξεκινήσει στους βασικούς τομείς υποστήριξης. αναφέρθηκε Καταρχάς το θέμα της ε, υποστήριξης ε, των πιο ευάλωτων προσφύγων. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο της υποστήριξής μας. Η δυνατότητα να προσφέρουμε στους πιο ευάλωτους που ανέρχονται σε 1,2 εκατομμύρια να λαμβάνουν ε, κάθε μήνα μετρητά Η διευκόλυνση αυτή υποστηρίζει τις οικογένειες ε, στην πρόσβαση στην εκπαίδευση με μια σειρά προγραμμάτων. Πέρα από την οικονομική υποστήριξη που παρέχεται, αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και αντιπροσωπεύει περίπου το μισό των τριών δισεκατομμυρίων που προσφέρουμε. Αποτελεί δηλαδή άμεση βοήθεια προς τις οικογένειες ε, στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. Όσον αφορά τη μη ανθρωπιστική πλευρά, το άλλο μισό των τριών δισεκατομμυρίων διατίθεται κατόπιν στενής συνεργασίας με τις τουρκικές αρχές και τους άλλους εταίρους μας. Αφενός για την εκπαίδευση, και εδώ είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι υποστηρίζουμε το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα, από τον υπηαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Η πρόκληση είναι να αποφύγουμε μια χαμένη γενιά όσον αφορά την εκπαίδευση. Επίσης, προσφέρουμε εξοπλισμό. Θα εξοπλίσουμε 125 σχολεία μόνιμης εγκατάστασης ε, και 50 σχολείων προκάτ. Σύντομα θα εκδώσουμε την ε, δεύτερη ετήσια έκθεση σχετικά με αυτήν την ε, διευκόλυνση. Στις 7 Μαρτίου θα δοθεί στο Κοινοβούλιο. Να σας δώσω και κάποια άλλα αντικειμενικά στοιχεία. Όσον αφορά την εκπαίδευση, υποστηρίξαμε την εκμάθηση τουρκικής γλώσσας για πάνω από 300.000 παιδιά. Δώσαμε μισθούς για πάνω από 5.000 ε, Τούρκους καθηγητές γλώσσας. Αναφέρθηκα και στην ανώτατη εκπαίδευση. 43.000 φοιτητές ωφελούνται από σχετική κατάρτιση και πάνω από 30.000 παιδιά ε, ε, ε, έχουν μεταφορά προς τα σχολεία τους. Έτσι λοιπόν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση. Είδαμε διπλασιασμό εγγραφών ε, στα προγράμματα αυτά από τότε που αρχίσαμε τη συνεργασία μας ε, με την Τουρκία πριν από δύο χρόνια. Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουν εγκαθιδρυθεί διάφορα κέντρα υγείας σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές. Είχαμε πλήρη εμβολιασμό 217.000 ε, βρεφών και 760.000 ε, ιατρικές επισκέψεις έχουν πραγματοποιηθεί. Ραντεβού με τους γιατρούς. Όχι μόνο δηλαδή προσφέρουμε χρήματα, αλλά καταφέρουμε να ε, φτάσουμε, να έρθουμε σε επαφή με τους πιο ευάλωτους πρόσφυγες στην Τουρκία. Αυτή ήταν η πρόκληση που αντιμετωπίζαμε στην αρχή. Το 93% του πληθυσμού βρισκόταν εκτός καταβλισμών σε όλη τη χώρα. Πολύ σημαντικό στοιχείο λοιπόν της προσέγγισής μας είναι να λάβουμε υπόψη μας και τις κοινότητες υποδοχής που δέχονται την πίεση στα κοινωνικά του συστήματα σε τοπικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ξεκινήσαμε και θα θέλαμε να κάνουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Πιθανότατα να το καταφέρουμε αυτό με τη δεύτερη δόση της διευκόλυνσης. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη απόφαση. Είναι κάτι πάνω στο οποίο εργαζόμαστε ακόμα. Υπάρχουν ε, όμως οι προσδοκίες ε, στο πλαίσιο της δήλωσης του Μαρτίου του 2016 μετά την εξάντληση των τριών δισεκατομμυρίων να ανταποκριθούμε στην ε, δέσμευσή μας να ε, διαθέσουμε άλλα τρία δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η δουλειά που κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν με βάση την πρώτη δόση, αλλά θέλουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα με βάση την δεύτερη όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική ένταξη των προσφύγων. Η Αναμπέλ Ρόιγ αναφέρθηκε στους πρόσφυγες που ήδη έχουν λάβει άδεια εργασίας. Χρειάζεται λοιπόν μια σφαιρική προσέγγιση, μια ολιστική προσέγγιση. Ήδη έχουμε ανθρώπους ε, που εργάζονται πάνω στις δεξιότητες ε, των προσφύγων, τις γνώσεις τους όσον αφορά τη γλώσσα. Αυτό είναι κάτι ε, το οποίο θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές. Θα θέλαμε επίσης να αναπτύξουμε το επιχειρηματικό πνεύμα αυτού του πολύ δραστήριου συχνά τμήματος του πληθυσμού. Η επίσημη αριθμή είναι μόλις η κορυφή του παγόβουνου. Θα δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να γίνει πιο ορατή η οικονομική συνεισφορά τους στην τουρκική κοινότητα. Την τουρκική κοινωνία, συγγνώμη. Αυτά είχα να πω λοιπόν κυρίως. Όσον αφορά τις υποδομές, να αναφέρω ότι στην υγεία Έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες για δύο νοσοκομεία, ώστε να έχουμε και πιο μακροπρόθεσμη διαρθρωτική υποστήριξη προς την Τουρκία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Έχετε το λόγο κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Αλλά είναι πάρα πολύ επιβαρημένη η κυκλοφορία 4 με 4,5. Και δύσκολο είναι να είναι κανείς ο τελευταίος ομιλητής, διότι πολλά ελέγχθησαν και ελπίζω ότι δεν θα επαναλάβω κάποια θέματα τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί. Πάρα πολύ σύντομα θα σας αναφέρω κάποιους αριθμούς. Μιλούμε για 3,5 εκατομμύρια Συρίους. 1,8 τα οποία είναι παιδιά. Είναι σημαντικός αυτός ο αριθμός. Και πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για έναν αριθμό που ξεπερνάει τον πληθυσμό 7 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι κάποιοι δεν ε, συνειδητοποιούν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα αυτό. Επίσης, Έχουμε περίπου 320.000 Ιρακινούς, ε, υπόλοιπους Ασιάτες, Αφγανούς, που επίσης έχουν ζητήσει άσυλο στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν είναι η μεγαλύτερη χώρα φιλοξενίας προσφύγων και τον άσυλο στον κόσμο. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Βρίσκονται παντού. Δεν του κρατούμε σε κέντρα, σε στρατόπεδα, σε καταβλισμούς. Όπως ελέγχθη, περισσότερο από 94% των Συρίων συμβιώνουν με τους Τούρκους. Μοιραζόμαστε σπίτια, κέντρα υγείας, σχολεία και μέχρι τώρα το κράτος, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν δαπανίσει περισσότερα από 30 δις. Όλο και περισσότερο αυξάνεται το αριθμό τα τελευταία χρόνια αν κάνετε συγκρίση με την αρχή της κρίσης. Βρισκόμαστε στο 7ο έτος της κρίσης αυτής. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στις πόλεις. Αν πάει καλή στο Χατάι, ένα τρίτο του πληθυσμού προέρχεται από τη Συρία. Στο, στο Γκαζιαντέπ το 1 τέταρτο. Το Γκαζιαντέπ είναι ε, πόλη, έχει 2 εκατομμύρια κατοίκους. Έχετε λοιπόν 500.000 Συρίους στο Γκαζιαντέπ και υπάρχει η επαρχία της Κιλής όπου Υπάρχουν περισσότεροι Σύριοι από Τούρκοι, αν θέλετε. Δηλαδή, έχουμε 110.000 Συρίους, 100.000 Τούρκους. Αν δείτε τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, περίπου έχετε 550.000 που ζουν εκεί. Βρίσκονται παντού δηλαδή. Αν δείτε πόσους φοιτητές από τη Συρία έχουμε. Σήμερα έχουμε περίπου 610.000. Δημιουργούμε σχολεία στους, ε, στα κέντρα στα οποία ε, μένουν για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες και βεβαίως δεν μιλούμε μόνο για πρόσφυγες από τη Συρία, πρέπει να μιλήσουμε και για τους Συρίους οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Τουρκία. Έχουμε 208.000 μωρά που γεννήθηκαν στην Τουρκία και όλο και περισσότερο 280.000 με συγχωρείτε και ακόμη περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός τους. Παιδιά λοιπόν, μωρά που έχουν γεννηθεί στην Τουρκία. Επίσης, στα νοσοκομεία μας έχουν νοσηλευθεί και εγχειριστεί περισσότερο από ένα εκατομμύριο Σύριοι. Αυτή είναι η αριθμή. Και θα ήθελα να επιφερθώ τις ευκαιρίες που μου δίδεται για να αναφέρω πώς προχωρεί η συμφωνία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστατικό και το προσφυγικό. Δεν ε, γίνονται πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που όλοι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λειτουργεί λοιπόν το σύστημα. Έτσι με τον τρόπο αυτό έχουν μειωθεί και οι ε, παράνομοι ε, πρόσφυγες οι οποίοι φεύγουν από την ε, Τουρκία και πηγαίνουν στην Ελλάδα. Πρόκειται λοιπόν για μεγάλη επιτυχία και βεβαίως αυτό ε, μας οδηγεί στο να μην έχουμε και τους θανάτους που είχαμε στο Αιγαίο. Είχαμε πέρσι πολλές χιλιάδες θανάτους στην Αιγαίο. Επίσης, το λαθρεμπόριο κατά των προσφύγων είναι κάτι το οποίο επίσης έχει περιοριστεί. Όσον αφορά την εφαρμογή. Κράτησε τις υποσχέσεις της η Ευρωπαϊκή Ένωση για την συμφωνία ένα προς ένα. Έχουν ε, από τα ελληνικά νησιά επανέλθει 2.200 άτομα τα οποία σύμφωνα με τις συμφωνίες μπορούν να επανέλθουν και περίπου 12.200 έχουν αποσταλεί βάσει αυτής της συμφωνίας. Άρα έχει κρατήσει τις ε, συμφωνίες και τις υποσχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε προβλήματα τώρα. Τι μας είχε υποσχεθεί επίσης ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι θα επιταχυνθεί το ποσό των τριών εκατομμύριων που έπρεπε να δοθούν όχι στην Τουρκία, αλλά στους πρόσφυγες του Συρίου στην Τουρκία. Τα χρήματα λοιπόν δεν ε, παίρνει τα χρήματα τον εαυτό της, αλλά τρία θεσμικά όργανα παίρνουν αυτά τα χρήματα πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτά τα δήματα χορηγούνται στους Συρίους που είναι στην Τουρκία. Από αυτά τα τρία δις λοιπόν, σωστά είπε ο Πάτρικ, ότι έχουν χορηγηθεί και δαπανηθεί για τους Συρίους, αλλά βεβαίως πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα το 1,9 δις έχει δοθεί στους Συρίους, τα άλλα, ε, το υπόλοιπο 1,1 έχει δεσμευθεί και θα δοθεί τους επόμενους μήνες. Θα θέλαμε να επιταχύνει την όλη διαδικασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτό το θέμα. Από την άποψή τη έχουν δαπανηθεί τα χρήματα αυτά. Τα κράτη-μέρη λοιπόν, όπω υποσχέθηκαν, θα πρέπει να επιταχύνουν την ε, διαδικασία της δεύτερου ε, ποσού των τριών δις το οποίο πρέπει να φτάσει επίσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουν οι εργοί κρατών και κυβερνήσεων σύντομα. Παρακαλώ, θα ήθελα να ακούσετε αυτή τη σύγκριση που θέλω να κάνω τώρα. Μιλούμε για 30 δις τα οποία έχουν δαπανίσει οι Τούρκοι. Τι σημαίνει αυτό. Ο καθένας ίσως 385 ευρώ. Ο μέσος Τούρκος Δηλαδή καταβάλει ως υποστήριξη του Συρίου 385 ευρώ ο καθένας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμεύσει, έχει εν μέρη δαπανίσει, τρία δις όπως είπαμε, και αν κάνετε τον υπολογισμό με τον πληθυσμό των κρατών ε, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανίσει 6 ευρώ σε δύο χρόνια ανακάτοικο. Ενώ εμεί 385 επαναλαμβάνω. Αυτά είναι τα χρήματα που δαπάνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο τελευταία χρόνια. Έξι περίπου ευρώ. Αλλά βεβαίως Θα πρέπει ίσω να γίνουν κάποιε μικροδιορθώσει στου αριθμού που δίνουν, αλλά υπάρχει όπω καταλαβαίνετε μία πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και βεβαίω και το ΑΕΠ και το μέσο όρο ζωή στην Τουρκία είναι πολύ χαμηλότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει λοιπόν, πρέπει να πω, γίνει μεγάλη θυσία εκ μέρου του τουρκικού λαού για να βοηθηθούν οι πρόσφυγε, κυρίω οι Σύριοι. Γι' αυτό θα θέλαμε τα επόμενα τρία δις να διατεθούν το συντομότερο δυνατό. Επίσης, υπάρχει μια υπόσχεση την οποία δεν έχει κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η εθελού, το εθελούσιο πρόγραμμα ε, επιστροφής. Είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα με νόμιμο τρόπο μέσω του προγράμματος ανθρωπιστικής εθελούσιας εναλλαγής. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει γίνει. Βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι θα προχωρήσει σύντομα. Δεν ξέρω βεβαίως, η αριθμή δεν είναι τόσο σημαντική. Δεν ξέρω πόσοι Σύριοι θα ήθελα να πάρουν σε νόμιμα, σε εθελούσια βάση χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει αυτή η δυνατότητα να παραμείνει ανοιχτή. Δεδομένου ότι του είπαμε ότι υπάρχει νόμιμος τρόπος να κατοικήσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην κινούνται παράνομα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ανοίξει αυτή η δυνατότητα δεδομένου ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις θεωρητικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει τώρα να γίνει αυτό συγκεκριμένο. ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα στο οποίο έχουμε συμφωνήσει. Δεν θα επαναλάβω πολλούς αριθμούς που έχουν ήδη προαναφερθεί, αλλά θα ήθελα να προσθέσω, όπως ανέφερε και ο Πατρίκ, καθώς και η συνάδελφος από τον ΟΗΕ, ότι με το δεύτερο ποσό, τη δεύτερη δόση των τριών δίσε θα εστιαστούμε σε τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα, τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δαπανηθούν για την ενσωμάτωση, για την ένταξη των Συρίων, διότι φαίνεται ότι οι σειράξει στην Συρία δεν θα ολοκληρωθούν ούτε σε μήνες ούτε σε χρόνια. Ακόμη και αν συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να δούμε τι μένει μετά, τι θα συμβεί μετά. Κοιτάξτε το Ιράκ. Τελείωσε ο πόλεμος πριν από πάρα πολλά χρόνια αλλά υπάρχουν ακόμη 200.000 ε, Ιρακινοί που ήρθαν ε, ως παράνομοι μετανάστες στην Τουρκία και ακόμη παραμένουν στη χώρα μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πραγματιστές. Υπάρχουν κάποια άτομα, τα παιδιά, οι φοιτητέ που χρειάζεται να τα εντάξουμε στις κοινωνίες μας. Για τα επόμενα λοιπόν αυτά τα τρία δις θα πρέπει να εστιαστούμε στην ενσωμάτωση, στην ένταξη. Πρώτο θέμα. Δεύτερο, κάποιοι από τους Σύριους άρχισαν να θέλουν να επανέρχουν, να ξαναγυρίσουν τη Συρία. Εκεί δεν είναι σταθερά τα πράγματα. Υπάρχουν άτομα τα οποία θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους διότι απελευθερώθηκαν από την ΤΑΕΣ και από άλλες δυνάμεις από την TID και στις περιοχές Αλμπάβ ε, έχουν επιστρέψει στην Τουρκία γύρω στα 100.000 άτομα σε αυτές τις περιοχές που προανέφερα. Στην επόμενη λοιπόν χρηματοδότηση που θα έχουμε θα πρέπει να εστιαστούμε και στο πώς θα δαπανίσουμε σωστά αυτά τα χρήματα. Τρίτη παρατηρησή, το στοιχείο που θέλω να τονίσω. Οι Δήμοι και οι κοινότητες. Ίσως κάποιοι από εσά ακούσατε τι είπε δήμαρχος Γκαζιαντέπ, η δήμαρχος του Γκαζιαντέπ πριν από ένα μήνα που είπε ότι στην πόλη της το 1 τέταρτο αποτελείται από Συρίους. Δηλαδή, μιλάμε για σχεδόν για το μισό πληθυσμό των Βρυξελών. Και είπε ότι Γι' αυτό αναφέρω ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στις διάφορες Δήμου και κοινότητε στι διάφορες πόλεις, στι διάφορες περιοχές. Μέχρι τώρα τρία ε, υπουργεία τουρκικά, άλλα θεσμικά όργανα, φορείς ε, και ΜΚΟs ασχολούνται με αυτά τα θέματα, αλλά θα πρέπει να συμμετάσχουν στο όλο εγχείρημα και οι δήμοι και οι κοινότητες που είναι κοντά στα άτομα. Γνωρίζουν εκ του σύνεγγυς τα προβλήματα που έχουν οι πρόσφυγες μετανάστες και θα πρέπει να τους εντάξουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλουμε. Όλα αυτά τα λέγω για να πω πού θα ε, στοχεύσουμε με τα δεύτερη δόση αυτών των τριών δις που περιμένουμε. διότι όντως επιτόπου στα διάφορα μέρη χρειάζονται αρρωγή και βοήθεια μεγάλη τα άτομα αυτά. Επίση ε, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το τι διαμείβεται αυτή τη στιγμή στο Αφρίν. Ξέρω ότι πολλοί πιστεύουν ότι και εκεί έχει πολλούς πρόσφυγες, αλλά είδαμε τι έγινε στην επιχείρηση που αναπτύχθηκε κοντά στην περιοχή του Εφράτη αυτή υπήρξαν εσωτερικές μετακινήσεις και έχουμε ε, περισσότερους από 130.000 Σύρους οι οποίοι έχουν πάει στις πόλεις που προανέφερα. Όταν λοιπόν απελευθερωθεί από τις τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η DOS, η PUID το Αφρίν, ελπίζουμε ότι τουλάχιστον 300.000 ε, θα μπορέσουν να μετακινηθούν εκεί. Οι μισοί, τουλάχιστον 350, βρίσκονται στην Τουρκία. Δεν μπορούν σήμερα να επιστρέψουν στη χώρα τους, δεδομένου ότι υπάρχει το PID και το YPG. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να επανέλθουν στην περιοχή τους, στην περιοχή της επαρχίας του Αφρίν, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που προανέφερα. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι θα επιληθεί το πρόβλημα του επόμενου μήνες. Ε, the Ευχαριστούμε τον κύριο Πρέσβη. Τα μέλη τώρα έχουν το λόγο, παρακαλώ. Ja ε, vielen Dank. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους και, εγώ και ο κύριος Πρέσβης ήρθαμε αργά λόγω της συμφόρησης στην πόλη και δυστυχώς ε, έχασα ένα κομμάτι από τις παρουσιάσεις. Άκουσα όμως και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι από την παρουσίαση του κυρίου Πακέτ. Ένα ερώτημα έχω προς τον κύριο Πρέσβη. Ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο στο θέμα της εκπαίδευσης. Είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό. Ο κύριος Πακέτ το είπε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρξει μια χαμένη γενιά για, από τους ε, πρόσφυγες. Οι, πρόσφυγες, οι άνθρωποι αυτοί είναι σημαντικοί. Γιατί αυτοί θα χτίσουν ξανά από τα συντρίμια τη χώρα τους. Και σωστό ε, είναι να λάβουν εκπαίδευση. Αλλά ε, εδώ και κάποιες εβδομάδες, ήδη από τα τέλη του προηγούμενου έτους, αποφασίστηκε από την τουρκική κυβέρνηση ότι τα συριακά σχολεία για τα παιδιά των Σύρων θα κλείσουν παρόλο που χτίστηκαν από τους Σύρους και ότι τα παιδιά θα πάνε σε τουρκικά σχολεία. Υπάρχουν και μαθήματα τουρκικής γλώσσας. Σωστό είναι αυτό, τα παιδιά οι νέοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν στην Τουρκία, αλλά φυσικά δεν είναι γνωστό πότε θα μπορέσει κανείς να επιστρέψει στη χώρα του. Αλλά το ερώτημα είναι, αν όντως επιστρέψουν στη χώρα τους, και έχουν μάθει τουρκικά και ε, ίσως δεν ξέρουν ή δεν μαθαίνουν πια τα αραβικά, τη μικτρική τους γλώσσα δηλαδή, θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω στη Συρία κάποια στιγμή και να μπορέσουν να βοηθήσουν στην ε, ανοικοδόμηση της χώρας. Ή αυτή η ένταξη που γίνεται ήδη τώρα, και δεν το εννοώ αρνητικά, Μήπως αποτελεί ένα μέρος ενσωμάτωσης ε, για να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι Τούρκοι πολίτες ας πούμε. Φυσικά το μέλλον είναι εντελώς αβέβαιο, αλλά το ερώτημα νομίζω ότι πρέπει να το θέσουμε. Εγώ είμαι από τη Γερμανία και σε εμά υπάρχουν ε, ε, μαθήματα μητρικής γλώσσας και για παιδιά Τούρκων. Γι' αυτό το σκέφτομαι αυτό που σας ρωτώ. Οπότε φαντάζομαι πόσο δύσκολο, σχεδόν αδύνατο είναι και για εσάς να οργανώσετε μαθήματα αραβικής γλώσσας, αν το σκεφτούμε από απλά οικονομική πλευρά για τα παιδιά των προσφύγων. Αλλά δεν θα ήταν αυτό πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό δεν θα μπορούσαμε κάποια κομμάτια αυτή τη δεύτερη δόση του Ευρωπαϊκού Κονδυλίου να τα χρησιμοποιήσουμε για το σκοπό αυτό. Και επίση άλλο ένα ερώτημα. Με τους σύρους δασκάλου καθηγητέ, τι γίνεται. Αυτούς δηλαδή που μέχρι τώρα δούλευαν, δίδασκαν στα σύριακα σχολεία στην Τουρκία και δίδασκαν τα παιδιά των σύρων προσφύγων. Για αυτούς τι δυνατότητες υπάρχουν θα ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της ε, Τουρκίας και θα διδάσκουν εκεί. Και μετά, ε, σημείωσε κάποια αριθμητικά στοιχεία. 610.000 είπατε φοιτητές από την ε, Συρία υπάρχουν και επίσης πάρα πολλοί μαθητές, πολλά παιδιά βεβαίως μεταξύ των ε, Σύρων προσφύγων. Στην Τουρκία πώς το διαχειρίζεστε αυτό, γιατί πολλοί καθηγητές και πολλοί δάσκαλοι έχουν απολυθεί. Θα ξαναπροσληφθούν τι γίνεται με το προσωπικό δηλαδή που θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας. Μπορείτε να το εγγυηθείτε ότι υπάρχει. Και κάτι άλλο, ένα λεπτό. Όχι, αυτό ήταν το βασικό που θέλω να ρωτήσω. Και γενικώ ε, μπορεί κανείς να υπογραμμίσει και συχνά το κάνουμε και στο παρελθόν, αλλά και σήμερα θα το κάνω, ότι πραγματικά είναι σημαντική η προσφορά της ε, Τουρκίας στην διαχείριση, την αντιμετώπιση αυτής της απίστευτης κρίσης ε, και των μεγάλων όγκων προσφύγων. Ελπίζω όντως και εγώ τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν όντως, ε, να εγκρίνουν όντως άμεσα τη δεύτερη δόση του δανείου. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Σπασίς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους εξαιρετικούς ομιλητές που πήραν το λόγο σήμερα. Όπως θα γνωρίζει και η κυρία Ματίας, ε, πρόσφατα επισκέφτηκα μαζί σας το Λίβανο. Και μεγάλη λύπη μου άκουσα πρόσφυγες από τη Συρία να λένε ότι το 1948 μετανάστευσαν οι γονείς τους το 1948 από το σημερινό Ισραήλ ε, και τώρα ξανά είναι πρόσφυγες οι ίδιοι. Είναι πολύ πιθανό μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων να μην επιστρέψουν ποτέ στη Συρία. Δυστυχώς. Είναι εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει υποδεχόμενοι 3,4 εκατομμύρια ε, προσφύγων. Η Ευρώπη δυστυχώς ε, κόλλησε, δίστασε όταν ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες. Εσείς όμως έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά και βγάζω το καπέλο μου για τις προσπάθειές σας. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως περιγράψατε, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Η συγκεκριμένη μου ερώτηση είναι η εξής. Επιτρέπεται οι Σύριοι πρόσφυγες ε, να ανοίξουν επιχειρήσεις, διότι κάπου διάβασα ότι Σύρος Μιλισοκόμος στο Ιράκ έλαβε τα εργαλεία για να αποκτήσει πάλι μελίσια και να έχει εισόδημα και να φροντίσει την οικογένειά του. Αυτό είναι δυνατόν στην Τουρκία. Υπάρχουν χρήματα δηλαδή για να δημιουργήσουν επιχειρήσεις οι πρόσφυγες. Η δεύτερη μου ερώτηση. Είπατε, τα δύο τρίτα των προσφύγων είναι γυναίκες και παιδιά. Προβλέπετε μικροχρηματοδότηση για να μπορέσουν να φροντίσουν οι ίδιες την οικογένειά τους. Υπάρχουν μετρητά διαθέσιμα, διότι οι ίδιοι οι πρόσφυγες γνωρίζουν καλύτερα τι ανάγκες έχουν. Μπορεί να τους δίνουμε κουβέρτες και να μην χρειάζονται κουβέρτες. Χρειάζονται λοιπόν μετρητά για να αποφασίσουν οι ίδιοι τι χρειάζονται περισσότερο οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Η τρίτη μου ερώτηση είναι η εξής. Όσον αφορά την επανεγκατάσταση, νομίζω ότι είναι ηθικά σωστό η Ευρώπη να δείξει το ήθος της στους πρόσφυγες. Η Τουρκία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, υποδεχόμενη 3,4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Θα πρέπει και εμείς να συμμετάσχουμε στην επανεγκατάσταση κάποιων από τους πρόσφυγες στις χώρες μας για να επιδείξουμε την αλληλεγγύη μας στην Τουρκία και στους πρόσφυγες αυτούς. Τελευταία μου ερώτηση. Δεν υπήρχε κάποια διευκόλυνση όσον αφορά τις θεωρήσεις προς Τούρκους υπηκόους για την Ευρώπη στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και τέθηκε σε ισχύ αυτό ή όχι. Η κυρία Βόζεμπεργκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσαν σήμερα. Ε, ξέρετε ότι οι διεθνείς οργανισμοί, ε, έρευνες που έχουν γίνει από τους διεθνείς οργανισμούς, έχουν δείξει ότι αυτό το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Ματίας, ότι η προστασία που ζητείται από τους πρόσφυγες δεν είναι ε, αντίστοιχη με εκείνη την, η οποία ορίζεται από τη συνθήκη της Γενέβης, παρέχεται μια προσωρινή προστασία, σύμφωνα με την οποία όμως δεν διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως επιβάλλει η συνθήκη της Γενέβης, με πολύ σημαντικές ελλείψεις που ήδη έχουν αναφερθεί και στις εισηγήσεις σας και εξηγούνται με έναν τρόπο. Αυτό δείχνει μια δυσαρμονία του δικαίου έτσι όπως επιβάλλεται με εκείνο που ενδεχομένως θα ήταν το αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση, ε, ήδη μας ενημερώσατε ότι υπάρχει και μια, σε σχέση με τους σύρους πρόσφυγες, ανεπαρκής πρόσβαση στην εργασία, είτε διότι ε, δεν υπάρχει δυνατότητα της επαρκούς εκπαίδευσης και γνώσης της γλώσσας, είτε έχει να κάνει ενδεχομένως με ειδικότητε που δεν μπορούν να καλυφθούν. Ε, ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Ήδη έχει καταγραφεί και εσείς κύριε Πρέσβη εστιάσατε περισσότερο στο κατά πόσον οι οικονομικοί πόροι που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επαρκείς και στον τρόπο με τον οποίο δίνονται ούτως ώστε να απορροφηθούν από την Τουρκία σχετικά με τα προγράμματα στα οποία αναφέρονται οι πόροι αυτοί. Ε, την κατάσταση τη γνωρίζουμε. Εγώ ήθελα να ε, σας θέσω ουσιαστικά ένα ερώτημα που δεν αναφέρθηκε, δεν είδα να αναφερθείτε. Αναφερθήκατε στις ευάλωτες ομάδες, αναφερθήκατε στα παιδιά και το κατά πόσο υπάρχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και πώς ε, ε, κατοχυρώνονται τα δικαιώματά τους. Το ένα μου ερώτημα είναι πώς σκέφτεστε να καλυφθεί το κενό της διαφοράς του προστασία της προστασίας που παρέχεται από την οφειλόμενη προστασία με βάση τις συνθήκες της Γενέβης. Το δεύτερο και που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι αν έχετε καταλήξει ποιος είναι ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων και τι ακριβώς ε, πρόβλεψη υπάρχει για τη διαχείριση αυτού του πολύ ευαίσθητου και εξειδικευμένου τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you so much. Uh, Mrs. I'm sorry. Ευχαριστώ η κυρία Σόιντροβα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ τις προσπάθειες που καταβάλλονται υπέρ των προσφύγων. Και αυτό το οποίο γίνεται στην Τουρκία. Δύο ερωτήσεις έχω να σας υποβάλω μιλήσατε για τους κανονισμούς που αφορούν την προσωρινή προστασία. Τι εννοείτε χρονικά όταν λέτε προσωρινά. Σε χρόνια Φερρυπίν. Το εκτιμώ ως μέσον που χρησιμοποιείτε, ως νόμιμο μέσον, αλλά ποια είναι η χρονική διάρκεια αυτού του μέσου. Δεύτερον, όσον αφορά την παιδεία, την εκπαίδευση. Αναφέρατε ότι 1,5 εκατομμύριο παιδιά υπάρχουν εκεί. 38% είναι εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Έχετε κάποιο τρόπο να διευθετήσετε το θέμα αυτό, διότι πιστεύω ότι είναι πρωταρχική σημασία για το μέλλον των ατόμων και συγκεκριμένα αυτών των παιδιών το θέμα της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ κύριος Κύρκος. Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω και εγώ τους πολύ σημαντικούς ομιλητές. Ευγνώμονες για την Τουρκία, όπως ευγνώμονες και για το Λίβανο, ευγνώμονες και για την Ιορδανία. Εκατομμύρια προσφύγων έχουν βρει σπίτι σε αυτές τις χώρες ένας πολύ μικρότερος αριθμός βρήκε στην Ήπειρό μας και κόντεψε να μας γκρεμίσει. Δεύτερο, πολύ σημαντική η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπως είπε ο κύριος πρεσβευτής, και μόνο να σκεφτούμε ότι 12.000 Σύριοι μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη με τη συμφωνία 1 προς 1, ενώ μόνο 13.000 από τη μεγάλη μας προσπάθεια για το resettlement. Βλέπουμε δηλαδή πως οι αριθμοί είναι σχεδόν ίδιοι. Άρα είναι πολύ σημαντικό ως τρόπος. Στην αρχή η τουρκική θέση για τους Σύρους πρόσφυγες ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά. Βλέπουμε μέσα στο χρόνο πως η ρητορική για επιστροφή των Σύρων στη Συρία βαθαίνει και πως βλέπουμε και κυρίως στα αστικά κέντρα αυξάνει, ε, αυξάνουν τα περιστατικά βίας μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων. Είχαμε 2017 34 πρόσφυγες νεκρούς, των οποίων 24 ήταν Σύροι. Αυτό είναι κάτι που το κράτος πρέπει να το λάβει υπόψη. Μιλάμε για την αγορά εργασία. και λέμε πω μόνο 25.000 Σύριοι έχουν πάρει άδεια εργασία, Μα είναι φανερό από το 1 εκατομμύριο άνδρε οι οποίοι είναι α πούμε ικανοί για εργασία, το 25.000 είναι απίστευτα μικρό. Αλλά την ίδια στιγμή η παράνομη εργασία και για του ίδιου του Τούρκου είναι πάρα πολύ μεγάλη, σχεδόν το 1 τρίτο αν παρακολουθώ σωστά τι έρευνε. Άρα δεν δείχνει ότι ειδικά οι Σύριοι έχουν αυτό το πρόβλημα, πρέπει να ληφθούν θετικά μέτρα είτε με, τα, με, τα, ποσοστά, είτε με την ε, ε, περαιτέρω εκπαίδευση σε ικανότητες, αλλά να καταλάβουμε πως είναι ένα βαθύ πρόβλημα της ίδιας λειτουργικής οικονομίας. Για την εκπαίδευση όλοι θέλουμε και ελπίζουμε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ειδικά για τα παιδιά των προσφύγων που μιλάμε τώρα και για αυτούς τους πληθυσμούς ως Ευρωπαίοι πρέπει να καταλαβαίνουμε κιόλας πως η ριζοσπαστικοποίηση ενδεχομένω των νέων μπορεί να περάσει και από τη μη ένταξή του και στο σχολικό περιβάλλον και μετέπειτα στην οικονομία. Άρα πρέπει ακόμα περισσότερο να έχουμε στραμμένη την προσοχή μα πώ θα βοηθήσουμε την Τουρκία και αυτά τα παιδιά. Από την Τουρκία θα μπορούσα να συνοψίσω ό,τι ζητάμε. Χρηματοδότηση των Δήμων όχι με τη βάση του αριθμού των Τούρκων που έχουν, γιατί διάβασα πω έτσι γίνεται η επίσημη χρηματοδότηση, αλλά με τη βάση των κατοίκων, όπως μας είπε ο κύριος Καϊμαξή, πολλές φορές ξεπερνούν τους ίδιους τους Τούρκους και επίσης σύνδεση των τοπικών αρχών και των τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων με τα προγράμματα βοήθειας των προσφύγων γιατί γνωρίζουμε πως μέσα στον αυξημένο συγκεντρωτισμό του το τουρκικό κράτος πολλές φορές ε, βάλει, βάζει τα ίδια προγράμματα παντού σε ένα παπούτσι χωράνε όλα τα πόδια. Πρέπει να περάσουμε από την χωρίς κριτήρια ανθρωπιστική βοήθεια όπως υπόθηκε και από έναν συνάδελφο σε στοχευμένη βοήθεια σε μια κατεύθυνση βιώσιμης ε, sustainable είναι η αγγλική λέξη ζωής ώστε να δούμε ε, το επόμενο βήμα που δεν είναι οι πρώτες ανάγκες είναι ανάγκες πληθυνών που θα μείνουν χρόνια, κάποια χρόνια σε αυτή τη θέση. Και βοήθεια και νομοθετική αλλά και τεχνική για σύρους να μπορέσουν να ανοίξουν τις δικές τους εταιρείε, τις μικρομεσαίες, τις ατομικές επιχειρήσεις. Αυτό να σας ενημερώσω, ούτε στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να το κάνουμε. Παλεύουμε με το τέρας γραφειοκρατίας, διότι οι Σύροι έχουν αυξημένη ικανότητα και θέληση να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά η γραφειοκρατία τους εμποδίζει. Πρέπει και η Τουρκία να βρει τρόπο να τους επιτρέψει νόμιμα αυτό. Το πέμπτο είναι το μήνυμα. Πριν από λίγες μέρες έγινε μια συγκέντρωση του ΑΚΑ Πάρτι στις Βρυξέλλες. Το μήνυμα ήταν είμαστε μουσουλμάνοι, είμαστε Τούρκοι. Εγώ θα ήθελα να το δω αυτό το μήνυμα στην Τουρκία προς τους Ήρους. Είμαστε μουσουλμάνοι, όλοι είστε αδερφοί μας. Η αγκαλιά μας συνεχίζει να είναι ανοιχτή. Αυτό το μήνυμα εκπεμπόμενο από τα κρατικά μέσα και από τα κρατικά χείλη θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να αναστρέψει αυτή την τάση που ανέφερα στην αρχή, την ενδοκινοτική βία. Τώρα τα δικά μας, τα ευρωπαϊκά. Φυσικά τα 3 δισεκατομμύρια της δεύτερης δόησης της βοήθειας προς τους Σύρους με τον τρόπο που είναι ευρωπαϊκός, όσο και αν ε, καμιά φορά φαίνεται δύσκολο και καταλαβαίνω τον κύριο Καϊμαξή, το ίδιο λέει και ο δικό μα υπουργό. Η βοήθεια πηγαίνει σε NGO και δεν πηγαίνει στο κράτο για να μπορέσει σοφά να την διανύμει. Καλά κάνει και πηγαίνει σε NGO, να υπάρχει απόλυτο έλεγχο, αλλά έτσι είναι ο ευρωπαϊκό τρόπο, συνεργαζόμαστε με όλου αυτού. Αλλά επιπλέον και χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει με κάποιο τρόπο, έστω μέσω των Δήμων, μέσω κοινών επιχειρήσεων, μικροεπενδυτικά εργαλεία, δεν ξέρω τι, είναι στο ζήτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει. Κάνουμε επενδύσει σε ανθρώπους, δεν δίνουμε ανθρωπιστική μόνο βοήθεια. Και φυσικά ε, Συγγνώμη, έχουμε και άλλους συναδέλφους που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Συγγνώμη που σας διακόπτω, λέει η κυρία Ματίας. Είναι πολύ σημαντικό, το Κοινοβούλιο παλεύει, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, η Κομισιόν ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Ευχαριστώ. Thank you, Chairwoman. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ματίας, η ερώτησή μου θα είναι πάρα πάρα πολύ σύντομη. Διότι έχω ε, επιφυλάξεις για τη συζήτηση αυτή, δεδομένου ότι συμβαίνουν άλλα πράγματα στη Συρία και στην ε, Ανατολική Μεσόγειο. Μία ένα ειδικό ερώτημα των πρέσβη. Αν μας αφορούν οι πρόσφυγες από τη Συρία. Θα πρέπει να μας απασχολούν όχι μόνο αυτοί που βρίσκονται ήδη στην Τουρκία, αλλά και αυτοί οι οποίοι υποχρεώνονται εκ των γεγονότων να πάνε στην Τουρκία. Το ε, Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το Σάββατο αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην Συρία να σταματήσουν αμέσως τους βομβαρδισμούς και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η τουρκική κυβέρνηση ήδη ανήγγειλε ότι θα συνεχίσει, διότι είπε ότι πρέπει να πολεμήσει κατά των τρομοκρατών, όπως την YPG. Οποιαδήποτε για τις ε, Δικέ μας προδιαγραφές και τι αμερικανικές δεν πρόκειται για τρομοκρατικέ οργανώσεις αυτές που αναφέρετε. Πιστεύετε ότι με αυτό που κάνετε βοηθάτε του πρόσφυγες ε, από την Συρία. Ευχαριστώ. Και εγώ. Είχα να κάνω δύο Ο κύριος Μαυρίδης έκανε τη μία. Αφορά την Αφρίν πολλούς μας απασχολεί το τι διαμείβεται εκεί. Όχι μόνο για το γεγονό ότι ίσω έτσι έχουμε περισσότερες προσφυγές μετά από αυτή τη σύγκρουση, αλλά διότι υπάρχει μονομερής επίθεση εκ μέρους της Τουρκίας. Βεβαίως υπάρχουν διεθνείς κανόνες και γιατί βάσει αυτών δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τρομοκρατική οργάνωση στην οποία γίνεται η επίθεση. Αυτό όμως δεν είναι το θέμα της συζήτησής μας και της συνάντησής μας, αλλά αναφέρετε κι εσείς ότι υπήρχαν και εκ μέρους σας κάποιες ανησυχίες και ερωτηματικά για το Αφρίν. Όντως υπάρχουν. Ερωτηματικά για το τι ακριβώς γίνεται στο Αφρίν. Αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Είπα στην αρχή κάτι, δεν είσαστε εδώ και θα το επαναλάβω. Βεβαίως δεν μπορούμε να δώσουμε μαθήματα για το πώς πρέπει να μεταχειρίζονται οι άλλοι στα πλαίσια αυτής της ανθρωπινικής κρίσης τους πρόσφυγες. Και βεβαίως δεν συμφωνώ ίσως με αυτά τα οποία γίνονται, πάντα μιλούμε για χρήματα, για πολιτικές και όχι για τα άτομα. Ξέρω ότι έχουν καταβληθεί υπεράθρωπες προσπάθειες μέσα του τουρκού λαού για να υποδεχθεί τους πρόσφυγες και ίσως δεν κάνουμε εμείς το ίδιο. Ξέρουμε όμως ότι και στο Λίβανο και στην Ορδανία Υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες επίσης. Ούτως ή άλλως, εσείς οι τρεις χώρες αυτές που προανέφερα έχετε υποδεχθεί πολύ περισσότερες πρόσφυγες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν είμαστε εδώ να σας δώσουμε μαθήματα. Με κανένα τρόπο. Θα σε ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη, που είστε παρόν. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για την καταστρατήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τους πρόσφυγες. Διότι μιλήσαμε για κονδύλια, για αριθμούς, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα μας απασχολούν όλος ιδιαίτερος. Τι κάνουν οι τουρκικές αρχές. Και βεβαίως και εκ μέρους Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής και εδώ έχουμε ερωτηματικά, αλλά τώρα απευθύνουμε σε εσά. Σας ευχαριστώ. Και σας δίνω το λόγο τώρα για να απαντήσετε στα ερωτήματα που τέθηκαν. Κοιτώ και από τις δύο πλευρές για να δω ποιος θέλει να αρχίσει πρώτος. I think most of the questions for... Νομίζω ότι οι περισσότερες ερωτήσεις ε, ήταν προς τον κύριο Πρέσβη, αλλά μπορώ να πω λίγα λόγια σχετικά με τα όσα ξέρω εγώ και τα όσα ίσως δεν ήταν αρκετά σαφή. Να απαντήσω καταρχάς σε αυτό που είπε ο κύριος Πρέσβης. Δεν θα ήθελα να ασκήσω πίεση στα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, καταβολή της χρηματοδότησης. 72 προγράμματα έχουμε, 3 δισεκατομμύρια ευρώ ε, ε, ε, αντιπροσωπεύουν και έχουμε προχρηματοδότηση, εκ των προτέρων χρηματοδότηση. Μέχρι στιγμής δηλαδή 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο λογιστικό μας σύστημα. Αυτά έχουν ήδη εκταμιευτεί. Τα υπόλοιπα 1,1 θα εκταμιευθούν ανάλογα με την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Μερικά από τα προγράμματα αυτά διαρκούν μήνες ή χρόνια. Έτσι λοιπόν απαιτούνται κάποια χρόνια μέχρι την τελική πληρωμή. Και γι' αυτό εκκρεμούν ακόμα 1,1 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών. Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω το σεβασμό να βγάλω το, καπέλο στα κράτη-μέλη που ε, διάθεσαν τα χρήματα αυτά πέρα από τις, ε, τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Ουσιαστικά ακολουθείται ο κανόνας ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στα 2, δισεκατομμύρια αυτά έχουν συμβάλει τα κράτη-μέλη ανάλογα με το ΑΕΠ τους. και έτσι μπορούμε να στηρίξουμε και το σύστημα προστασίας και ασύλου στην Τουρκία. Χρηματοδοτούμε λοιπόν ε, τις ε, χώρες, τους ε, τόπους μετανάστευσης επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για αυτού του τύπου την βοήθεια. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να αναφέρω έχει να κάνει με την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αυτήν. Το έχουμε σκεφτεί το θέμα αυτό και έχουμε προσπαθήσει να καλύψουμε όλες τις πλευρές, όλες τις στοιχές του θέματος αυτού. Μια οικογένεια μπορεί να χρειάζεται επιπλέον μετρητά. Μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσουμε κίνητρα για τα παιδιά να πάνε σχολείο. Μερικές φορές τα παιδιά χρειάζονται πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο κάποια βοήθεια και τέτοια προγράμματα χρηματοδοτούμε. Μερικές φορές χρειάζονται διδασκαλία στα τουρκικά, για παράδειγμα, της τουρκικής γλώσσας. Και, και τα μαθήματα στα αραβικά αποτελούν τμήμα των προγραμμάτων μας. Και επίσης ε, για κάποιες οικογένειες πρέπει να υπάρχει και μεταφορά προς τα σχολεία διότι μπορεί να βρίσκονται μακριά από τα σχολεία. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια ολιστική σφαιρική προσέγγιση και σιγά σιγά αυτό θα πρέπει να επιτρέψει και στα υπόλοιπα παιδιά να λαμβάνουν εκπαίδευση. Στον κύριο Μπασίρ. Θα ήθελα τέλος να απαντήσω ότι όσον αφορά αυτό το δίχτυ ασφαλείας που ανέφερα, που προσφέρει μετρητά στις οικογένειες, ε, αυτό γίνεται υπομορφή ηλεκτρονικής πληρωμής κάθε μήνα. Έχουμε εντοπίσει τις οικογένειες, τις συγκεκριμένε αυτές οικογένειες και συνήθως έχετε δίκιο. Οι γυναίκες των οικοκυριών αυτών λαμβάνουν τα χρήματα, διότι συνήθω γνωρίζουν καλύτερα ποιε είναι οι ανάγκε του νοικοκυριού. Αυτό λοιπόν αποτελεί τμήμα της φιλοσοφίας του προγράμματος αυτού. Να προσφέρει ε, δυνατότητες διαβίωσης ε, χρηματοδοτώντας τα νοικοκυριά. Ε, Δύο λόγια για κάποια από τα σχόλια που έγιναν. Συμφωνώ απολύτως με το όσα είπε ο κύριος Πασίρ για την ανάγκη επανεκατάστασης εντός της Ευρώπης αλλά και σε άλλες χώρες. Είναι όντως ε, δείγμα αλληλεγγύης προς την Τουρκία και προς τους ίδιους τους πρόσφυγες. Να σας δώσω κάποια στοιχεία εδώ. Πέρσι, 2017, είχαμε σχεδόν 15.000 άτομα που πελάθηκαν από την Τουρκία επανεγκαταστάθηκαν. Περίπου 12.000 ήταν Σύριοι. Αυτό καταφέραμε στα πλαίσια της επανεγκατάστασης. Περίπου τα ίδια αριθμητικά στοιχεία για το 2016 και αρκετά λιγότερα στα προηγούμενα χρόνια. Για το θέμα της εκπαίδευσης, συμφωνώ απολύτως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όντω πρέπει να είναι κοινέ οι προσπάθειε για τη μεγαλύτερη ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Υπάρχουν πολλέ δραστηριότητε, ε, ε, υποστήριξη των ε, μαθημάτων γλωσσών, τύπο βιβλίων, και γενικώ ε, δυνατότητες περισσότερη ένταξη. Δουλεύουμε πολύ στενά με το Υπουργείο εκπαίδευση, με το Υπουργείο Παιδείας της ε, Τουρκίας ε, για την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια αλλά και μεγαλύτερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να απαντήσω στην κυρία Βόζεμπεργκ για τα κενά που υπάρχουν με τη συνθήκη της Γενέβης. να ξεκαθαρίσουμε το εξή. Έχετε δίκιο. Υπάρχει όντως κενό μεταξύ της μεταχείρισης των προσφύγων στα πλαίσια της ε, συνθήκης της ε, Γενέβης και του προσωρινού καθεστώτος. Αλλά δεν είναι παράνομο το κενό αυτό. Είναι δύο διαφορετικά τα καθεστώτα που εφαρμόζονται σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Τα δικαιώματα της συνθήκης της Γενέβης ισχύουν για μεμονωμένο καθεστώς, ανά άτομο δηλαδή λαμβάνει το καθεστώς της, ε, του πρόσφυγα και από αυτή τη στιγμή το πάρει μπορεί να εξασφαλίσει τα δικαιώματα της συνθήκης της Γενέβης. Το προσωρινό καθεστώς προστασίας προσφέρεται συλλογικά, σε συλλογικές αφήξεις, σε μια ομάδα ατόμων χωρίς ε, διαχωρισμό μεταξύ των ατόμων που αποτελούν την ομάδα. Και αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε επίγουσες ε, συνθήκες. Γι' αυτό και τα δικαιώματα είναι λιγότερα, ας πούμε. Βεβαίως υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου που δίνει καθεστώς ε, ε, πρόσφυγα και υπάρχει και το αντίστοιχο καθεστώς που δίνει προσωρινή προστασία. Και εκεί είναι διαφορετικά τα δικαιώματα που μπορεί να απολαμβάνει ένας πρόσφυγας. Και στην Τουρκία λοιπόν τα δικαιώματα είναι διαφορετικά γιατί καλύπτουν διαφορετικά πλαίσια και καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρέσβη. Σύντομος και εγώ θα είμαι. Πολλά τα ερωτήματα. Κυρία Σόμερ, το θέμα της γλώσσας θέσατε. Έχουμε 78 εκατομμύρια Τούρκους, δεν χρειαζόμαστε περισσότερους. Προσπαθούμε λοιπόν βεβαίως να τους μάθουμε Τούρκοι, αλλά πρώτα απ' όλα τη μητρική τους γλώσσα. Στα κέντρα έχουμε σε 22 κέντρα έχουμε 85.000 ε, μαθητές. Ένα τρίτο λοιπόν βρίσκονται στα κέντρα, στα σχολεία, δεν έχουμε πρόβλημα. Και έχουμε 2.500 σύρους, δασκάλους που διδάσκουν τη γλώσσα, αλλά βεβαίως υπάρχουν και σχολεία παντού στις μεγάλες, πόρες, στις μεγάλες πόλεις, τις οποίες ανοίγουμε τις θύρες για τους μαθητές, για τα παιδιά των Σύρων. Δηλαδή, μπορούν να μάθουν και τη γλώσσα τους. Υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη πολλά κέντρα στα οποία μπορούν να προσφέρουν την εκμάθηση της αραβικής γλώσσας στα παιδιά που πηγαίνουν στα τουρκικά σχολεία. Δεν θέλουμε να ξεχάσουν την μετρική τους ε, γλώσσα, δεν θέλουμε να βρίσκονται στους δρόμους, θέλουν να πάνε στο σχολείο και να μάθουν γλώσσες. Καταλαβαίνετε ότι ε, υπάρχει και το θέμα το, της βίας για τα παιδιά ή των προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπίσουν και τα δικά μας τα παιδιά στους δρόμους και εκείνα. Θέλουμε λοιπόν να τους προστατεύσουμε από αυτά. Έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινά προγράμματα υπέρ της προστασίας των παιδιών. Αυτό απαντά στο δεύτερο, πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο. Οι άδειε εργασίες, η επιχειρηματικότητα. Ήδη έχουμε χορηγήσει περίπου 25.000 άδειε εργασία σε σύρους. Και υπάρχουν και πολλοί επιχειρηματίες, άνδρες και γυναίκες που φτάνουν από το Χαλέπι στον Καζιαντέπ και δημιουργούν τις δικές τους ε, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εργοστάσια. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε όμως ότι η Τουρκία είναι ένα από τα πιο ε, ε, ε, από τα πιο σημαντικά κράτη που έχουν υψηλή ανεργία μεταξύ των νέων και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιούργησε προβλήματα το 2016. Τώρα βελτιώνονται τα πράγματα, αλλά ενθαρρύνουμε και τους νέους σύρους να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μικροχρηματοδότηση είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Γίνονται οι καλύτερες δυνατές διευκολύνσεις επίσης για να απασχολούν όλο και περισσότερο σύροι και, και υπάρχει και κάποια ενθάρρυνση από πλευράς ηθικής προς τους Τούρκους για να απασχολούν ε, Σύρους. Η μετεκατάσταση είναι κάτι που αναφέρθηκε από πολλούς είναι πολύ σημαντική και η επανεγκατάσταση και η μετεκατάσταση. Η Ιταλία και η Ελλάδα ξέρουμε ότι φέρουν το μεγαλύτερο φορτίο. Η Γερμανία και η Σουηδία επίσης έχουν ε, κάνει μεγάλες προσπάθειες και άλλοι όμως θα πρέπει να τις βελτιώσουν. Ε, κάνουμε μία ε, συγκριτική ανάλυση μεταξύ των πιο σημαντικών θεμάτων για τα θέματα της μετανάστευσης και βεβαίως ελπίζουμε ότι με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη δική σας συνδρομή και ελπίζω με την δική σας υποστήριξη που θα χρειαστεί να ψηφίσετε να προχωρήσουμε. Τώρα, η προσωρινή προστασία. Τι σημαίνει. Δεν σημαίνει χρονικά περιορισμένη, διότι θα μπορεί κανείς ε, να έχει χέρι του καθεστώτος του πρόσφυγα ή της προσωρινής προστασίας. Στην πράξη όμως η προσωρινή προστασία δίδει τα ίδια δικαιώματα τα οποία έχουν οι νόμιμοι πρόσφυγες, οι Σύροι στην Τουρκία. Αλλά υπάρχουν κανονισμοί, κανόνες στα πλαίσια του ΟΗΕ. Ε, δεν σημαίνει ότι στην πράξη υπάρχουν μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τα δικαιώματά τους όμως ίσως επειδή χρησιμοποιείται διαφορετική ορολογία. Στην παιδεία, τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο ώστε να ενσωματώσουμε περισσότερους νέους στο σύστημα παιδείας. Και εγώ μπορώ να σας κάνω την ίδια ερώτηση. Εσείς, τα κράτη-μέλη, τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε για να υποστηρίξετε την Τουρκία, το Λίβανο, την Ιορδανία, το Ιράκ, χώρες στις οποίες υπάρχουν εκατομμύρια πρόσφυγες. Διότι είναι και θέμα χρημάτων. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας ανέφερα κάποια παραδείγματα και αριθμητικά. Είπα ότι ο κάθε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανά για τους πρόσφυγες στην Τουρκία 6 ευρώ, ενώ εμείς κατά είναι οι Τούρκοι 385 περίπου όπως προανέφερα. Θα πρέπει λοιπόν να ευρεθούν λύσεις. Συμφωνώ. Ο κύριος Κύρκος είπε ότι φτάνουν τα χρήματα στην Τουρκία. Μήπως δεν κατάλαβα σωστά. Για τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουν για τους πρόστιγες. Κύριε Μαυρίδη, για το Αφρίν. Οι επιχειρήσεις αυτές θα ε, σταματήσουν την παράνομη εισρωή μεταναστών και προσφύγων σε αυτή την περιοχή. Ξέρουμε ότι 130.000 Σύρι γύρισαν στην περιοχή τους και θα μπορέσουν να ζήσουν στην επαρχία της Αφρίν διότι έχουμε στην Τουρκία 350.000 στην ε, πλειοψηφία τους Σύρους θέλουν να επιστρέψουν αλλά η TID, η YPG που εμείς πιστεύουμε ότι είναι τρομοκράτες δεν τους το επιτρέπουν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όταν ε, πολεμήσουμε την ΤΑΕΣ και όλους αυτούς θα μπορέσουν να επιστρέψουν. Για μας το ΠΚΚ όπως και άλλες οργανώσεις που προανέφερα είναι τρομοκρατικές οργανώσεις και θέλουμε να προστατεύσουμε τον κόσμο από την δράση τους. Ένα τελευταίο ερώτημα από την Συμπρόεδρο. Αυτό το οποίο κάνουμε στην Αφρίν συνάδει με την ε, χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την προστασία από επιθέσεις. Ήδη πρέπει να πω ότι έχουμε ε, στην ε, Κιλής και στην Χατάη περίπου 100 θύματα μεταξύ των στρατιωτών και στην αρχή θανατώθηκε και άμαχος ε, πληθυσμός. Το TID, YPDG για μας είναι τρομοκρατικές οργανώσεις βρίσκονται σε άμεση σχέση με το ΠΚΚ, η ονομασία ίσως δεν έχει μεγάλη σημασία, το ότι προσπαθούν να επιτεθούν στους πολίτες μας και να αλλάξουν δημογραφικά την περιοχή του Αφρίν και να δημιουργήσουν κάποιες στρατιωτικές δυνάμεις που θα είναι κοντά στα σύνορά μας είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. 55% των κατοίκων του Αφρίν είναι Άραβες, 35% είναι Κουρδί, ενώ τώρα έχουν αυξηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Έχουμε και Σύρους. Δεν μπορείτε όμως να αλλάξετε τη δημογραφία μιας χώρας. Θέλουμε όλοι οι Σύριοι να μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Αναφέρατε την δήλωση της 8ης Μαρτίου είπατε ότι δεν σας ικανοποιεί. Είμαστε όμως ρεαλιστές. Έχουμε 3,5 εκατομμύρια Σύρους στην Τουρκία. Δεν ξέρω πόσους έχετε στη Γερμανία. 1,2. Το θέμα είναι ότι με τόσο υψηλό αριθμό προσφύγων δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τους παραδιοσυκούς κανόνες πάντα. Αν έχετε κάτι καλύτερο από την περίφημη δήλωση της ανταλλαγής 1 προς αν έχετε μια καλύτερη λύση να μας προτείνετε, να μας την προτείνετε. Αλλά πιστεύουμε ότι κάθε πρόσφυγας θα πρέπει να έχει πλήρη δικαιώματα. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε 3,5 εκατομμύρια σύρους στην Τουρκία. Πρέπει με επίγοντα τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Οποιαδήποτε συμφωνία δουλεύει προχωρά, λειτουργεί, είναι καλή. Αλλά να έχετε καλύτερη νήση, εάν οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μας πούν ότι θα πάρουμε όλου του πρόσφυγες εμεί στις χώρε μα ό,τι καλύτερο για μας. Έχει λυθεί το πρόβλημα. Εάν οι χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση μα πούνε, α βρούμε όλοι μαζί ένα πρόβλημα για του. Ήρου, έχει καλώ. Αλλά δεν ζούμε σε έναν ιδεατό κόσμο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, μοιραζόμαστε το ψωμί, το νερό που πίνουμε με του Ήρου πρόσφυγε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επίσης, αναφέρατε και καταστρατηγήσεις και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιών. Βεβαίω υπάρχουν και τέτοιου προβλήματα. Μπορεί να συμβεί αυτό. Προβλήματα με την παιδική παράνομη εργασία, αλλά μεταξύ αυτών των 3,5 εκατομμυρίων, επαναλαμβάνω, υπάρχουν προβλήματα. Στην Τουρκία προσπαθούμε να βοηθήσουμε παρά τις οικονομικές μας δυσκολίες. Συγχρόνως πρέπει να πολεμήσουμε τρεις πολύ διάσημες τρομοκρατικές οργανώσεις, άρα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το ερώτημα μου λοιπόν προς εσάς είναι, τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε εσείς ως κράτη-μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως σας είπα, τα πρώτα τρία δις έφτασαν σε δύο χρόνια. Τα δεύτερα ε, δόση, αν θέλετε, αυτών των τριών δις, πότε θα φτάσει, πόσο καιρό θα κάνει για να βοηθήσουμε τους Σύρους όσο πιο γρήγορα και όσο καλύτερα γίνουν τα πράγματα θα είναι καλύτερο προς το συμφέρον όλων μας. Διότι η ασφάλεια της Ευρώπης αρχίζει στα σύνορα της Τουρκίας. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να επιληθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι αρχίζει τώρα μόλις αυτή η συζήτηση, θα είχαμε και άλλα πολλά θέματα να πούμε. Θα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσουμε και τους διερμηνείς που έμειναν παραπάνω χρόνο. Παραμένει εκρεμής και συνεχίζεται η συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Δεν έχει τελειώσει και πάλι σας ευχαριστώ.